Καλημέρα σας. Good morning. Dear colleagues. Good morning everyone. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Να συνεχίσουμε τις εργασίες μας από εκεί που είχαμε μείνει. Είμαστε στο σημείο 14, στην ώρα των ψηφοφοριών, Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες για την περίοδο 2008 έως 2013. Εισηγητής, ο κύριος Μωράες, Δεν ξέρω αν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ εισηγητής. έγκριση σχεδίου σύσταση για δεύτερη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Θα ψηφίσουμε λοιπόν. γιατί δεν είναι παρόν ο κύριος Δεν ξέρω αν κάποιος ε, θέλει να λάβει το λόγο εξ ονοματός του. Παρακαλώ, κυρία Λάμπερτ. Θέλετε το λόγο. Απλώς να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι πρόκειται για τις αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους πρόσφυγες, ε, το οποίο, οι οποίες ταιριάζουν και με τον Οργανισμό για την ε, ε, Υποστήριξη για το Άσυλο. Τα έχουμε υποστηρίξει αυτά και επομένω η Επιτροπή θα υποστηρίξει την γνωμοδότηση του συναδέλφου κυρίου Μωράες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλώ εξ ονόματος ε, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ο κύριος Μωράες φυσικά είναι στην ομάδα μας. Να πω ότι αν υπάρχει οτιδήποτε που αφορά στο θέμα αυτό θα ασχοληθώ εγώ με αυτά εξ ονόματός του. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από την Προεδρία, ο κύριος Μπούρος. Ωραία. Να ψηφίσουμε. ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν έχετε την κάρτα σας. Ωραία. Θα μετρήσουμε μία ψήφο επιπλέον. Ωραία. 40 ψήφοι υπέρ, 5 κατά, καμία αποχή και μία ψήφος υπέρ επιπλέον, επομένως είναι 41 υπέρ η ψήφοι. Εγκρίνεται λοιπόν η γνωμοδότηση. Να ψηφίσουμε τώρα την έκθεση Λάμπερτ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Το ίδιο αποτέλεσμα, 40 ψήφοι υπέρ, 5 κατά, μία αποχή, 41 ή ψήφοι υπέρ. Ε, ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 16. Θέσπιση κοινού προγράμματος επανεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εισηγητής ο κύριος Ταβάρες. Δεν θα ψηφίσουμε και τις δύο μαζί, θα ψηφίσουμε μόνο το σημείο 16, λέει ο Πρόεδρος ψήφος προσανατολισμού για το σχέδιο γνωμοδότησης για τη θέσπιση κοινού προγράμματος επαναγκατάσταση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρχεται η ψηφοφορία, κύριε Ταβάρες, θέλετε το λόγο. Να πω μόνο ότι ψηφίζουμε μόνο την πρωτοβουλία, την έκθεση πρωτοβουλίας και από εκεί και πέρα την ε, συναπόφαση εργότερα, έτσι. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 19. Υπέρ. Against. It's adopted. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Συγγνώμη, ζητάει ζητάει πρόεδρος, 23. Υπέρ, κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία 24 τώρα. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25, κατά τμήματα κατόπιν αιτήματος του και πρώτο τμήμα, υπέρ. Ο κύριος Σταβάρης θέλει το λόγο, παρακαλώ. Ναι. Να εξηγήσω απλώς ότι, εξ όσων καταλαβαίνω εγώ, το θέμα είναι ότι είχαμε προβλέψει θρησκευτικές και εθνικές οργανώσεις στην τροπολογία του κυρίου Παπα-Νικολάου, συγγνώμη, στη συμβαστική τροπολογία, για να βοηθήσουμε την επαναγκατάσταση των προσφύγων. Και το αίτημα κατά τμήματα είναι να ψηφίσουμε πρώτα τους θρησκευτικού οργανισμούς και μετά τους εθνικούς οργανισμούς. Θα ήθελα να ζητήσω ξεχωριστή ψηφοφορία για θρησκευτικέ και κινητικού οργανισμού. Είναι προφορική η τροπολογία αυτή, γίνεται δεκτή. Αντί για religious and ethnical που ψηφίζουμε ξεχωριστά, religious and community organizations. Ελπίζουμε να είναι ευρύτερο αυτό. Είναι κάποιο κατά κύριε Πρόεδρε, δεν είμαστε βέβαιοι τι εννοείται με το community organizations. Ο κύριος Κάσμαν. Κύριε Πρόεδρε, να πω στην Επιτροπή ότι είχαμε ένα αντίστοιχο πρόβλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάποιες από τις ομάδες της άκρας δεξιάς ε, περιγράφονται ως community organizations. Νομίζω ότι μπαίνουμε λοιπόν σε ε, σκοτεινά μονοπάτια εδώ και καλό θα ήταν να είμαστε λίγο προσεκτικοί αν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα. Καταλαβαίνω το πνεύμα της τροπολογίας που θέλει να τα συμπεριλάβει όλα, αλλά καλύτερα θα ήταν να τα αντιμετωπίσουμε λίγο αργότερα. Εξ όσων κατάλαβα κύριε Ταβάρη, η προφορική τροπολογία δεν γίνεται δεκτή, υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις, επομένως θα την ψηφίσουμε όπως ε, έχει στη γραπτή πρόταση. Κύριε Μπουσουτήλ συμβιβαστικά. Μήπως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, Civil Society Organization. Μάλλον όχι, υπάρχουν αντιρρήσεις. Επειδή λοιπόν υπάρχουν στάσει, θα ψηφίσουμε όπως έχει η ψηφοφορία στο γραπτό κείμενο. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς υπέρ. Συγγνώμη, ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 17 κατά, καμία αποχή, επομένως εγκρίνεται. Κύριε Μισελ, συγγνώμη, νομίζω ότι καθυστέρησα, δεν δούλεψε και υπερψήφισα όμως. 29 λοιπόν υπέρ, 17 κατά. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 29 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 30 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 31 υπέρ, κατά. 32 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Παράγραφος 26. Έχουμε μία νέα προφορική τροφολογία του κύριου Ταβάρες. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Κατά πίπτη. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Η 35 καταπίπτει. 36 κατά εγκρίνεται. Κύριος Λαμπρινίδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μια προφορική τροπολογία στη συμβιβαστική τροπολογία 1 μετά από διαβουλεύσεις και με τον εισηγητή ο οποίος συμφωνεί με την τροπολογία, να προσθέσουμε στο τέλος της συμβιβαστικής τροπολογίας 1, η οποία αναφέρεται στην, ε, ε, στο ψήφισμα του 2001, το εξής. Implemented in the future per the Parliament's request. That's the oral amendment. Αυτή είναι η προφορική τροπολογία. Μπορείτε να την επαναλάβετε παρακαλώ. Such programs must also be implemented in the future per the Parliament's request. Any objection? Αντιρρήσεις. Ενστάσεις για την προφορική τροπολογία του κυρίου Λαμπρινίδη. Κύριε Κάσμαν, είστε αντίθετο? Είστε υπέρ. Ωραία λοιπόν. Ποιος είναι υπέρ λοιπόν. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα 38. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 40. Συγγνώμη, τη 39 ξέχασα. 39 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Από ό,τι βλέπω απορρίπτεται. 42. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Οι 43, 44 και 46 καταπίπτουν. υπολογία 45 θα πρέπει να ψηφιστεί. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται νομίζω. Τροπολογία 1. Για την προπομπή 5α νέα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. 9. Υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ εκτιμώντας α τροπολογία 3 υπέρ κατά νομίζω εγκρίνεται Τροπολογία προφορική του κυρίου Ταβάρες. Βλέπετε την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Αν και νομίζω ότι εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Όχι, εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Καταπίπτει. Θέλετε να τι ψηφίσουμε όλε μαζί. Όχι, δεν γίνεται δεκτό το αίτημα. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 17. 17. Πέραση ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 21 κατά, εγκρίνεται. 23 υπέρ, 22 κατά, εγκρίνεται. Και τροπολογία 18 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. 39 υπέρ, 4 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ κύριε Ταβάρας. Και τώρα να ψηφίσουμε το δεύτερο κείμενο και το σχέδιο έκθεσης. Κύριε Ταβάρες, θέλετε το λόγο. Let's go for the vote. Starting. Amendment 2 withdrawn. Τροπολογία 2 έχει αποσυρθεί. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 10, η 11, 12, 13, 14. Η 3 έχει αποσυρθεί. Η συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Καταπίπτει 15 και 16. 4. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Δεν χρειάζεται. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτηκε νομίζω. 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 1 κατά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Όχι. Εγκρίνεται. 9. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρο... Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. 39 υπέρ, 5 κατά, χωρίς αποχές. Πρόκειται λοιπόν για μια ψηφοφορία προσανατολισμού. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Σας ευχαριστώ. Και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 18. Πρόκειται για το δικαίωμα διερμηνίας και μετάφρασης σε ποινικέ διαδικασίες. Η κυρία Λάτφορτ κυρία Λάτφορτ είναι η συγγήτρια και εδώ πρόκειται για ψηφοφορία προσανατολισμού. Έχετε το λόγο κυρία Λάτφορτ. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν θέλω να καθυστερήσω την ψηφοφορία παραπάνω. Αλλά θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την συμμετοχή τους, την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε ήταν πάρα πάρα πολύ χρήσιμη. Και βλέπετε το αποτέλεσμα αυτής της επιτυχημένης συνεργασίας ότι υπάρχουν τόσο πολλές συμβαστικές τροπολογίες, 18. Πραγματικά είμαστε όλοι σύμφωνοι όσον αφορά τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές. Ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα τους συναδέλφους και ζητώ από όλους σήμερα να τη στηρίξουν. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά συν. Είναι οι συμβιβαστικές ε, τροπολογίες. Οι δικές μου τροπολογίες πολλές φορές καταπίπτουν, αλλά βλέπετε ότι είμαι υπέρ και έχω βάλει ένα συν δίπλα από τις περισσότερες τροπολογίες. Δύο σχόλια μόνο θέλω να κάνω. Πρώτον, στην τροπολογία 39 που είναι στον δεύτερο κατάλογο, εδώ υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Η τροπολογία 39 είναι για να μπει στο κείμενο της οδηγίας και όχι του νομοθετικού ψηφίσματος. Αυτό το σημείο θα μπορούσε άνετα να ενσωματωθεί στο νομοθετικό ψήφισμα. Και θα ήθελα πραγματικά να πω εδώ ότι όσον αφορά το περιεχόμενο, η πρόταση της Επιτροπής μπορεί να μας βρει σύμφωνος. Αλλά όπως είπα και στην συζήτηση που είχαμε, υπάρχουν κάποιες νομικές, αν θέλετε, περιπλοκές. Εάν παραθέσουμε εδώ το κείμενο της οδηγίας σε αυτό το νομοθετικό ψήφισμα. Προτείνω λοιπόν μια προφορική τροπολογία και αντί να πούμε εδώ ότι αναφερόμαστε στο κείμενο της Επιτροπής, να πούμε ότι λαμβάνουμε υπόψη μας το γεγονός ότι η Επιτροπή κάνει μία πρόταση. Αλλάζουμε λίγο την διατύπωση και ε, κατά κάποιο τρόπο κάνουμε μία διαφορετική αξιολόγηση αυτής της πρότασης. Και πραγματικά εκτιμούμε την εργασία που έγινε, αλλά ελπίζω εδώ να δείξετε κατανόηση, γιατί με αυτή τη νέα διατύπωση αποφεύγουμε αυτό που προηγουμένως ονόμασα νομικές ε, περιπλοκές που μπορεί να προκύψουν. Δηλαδή, ουσιαστικά αναφερόμαστε στην πρόταση της Επιτροπής, στην ουσία της, αλλά από διαδικαστικής απόψεως διατηρούμε τις ε, προϋποθέσεις που πρέπει κατά τα άλλα λοιπόν και εκτός από αυτήν την προφορική τροπολογία και με αυτόν τον τρόπο μπορώ να είμαι υπέρ της τροπολογίας 39. Ευχαριστώ πολύ και το ΕΛΚ που φαίνεται ότι μπορεί να δεχτεί αυτή την πρότασή μου. Άλλη διαφορά που συνεχίζει να υπάρχει είναι στην παράγραφο 6 και εδώ μιλάμε για τις προφορικές μεταφράσεις. Έχουμε την 84 του κυρίου Κοέλιο Και εδώ υπάρχει η τροπολογία του συναδέλφου μου, του κυρίου Άλβαρο. Συνεχίζω όμως εδώ να πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την τροπολογία 30. Δηλαδή υπάρχουν εδώ εγγυήσει όσον αφορά την προφορική τροπολογία. Ενδυναμώνουμε δηλαδή αυτές τις εγγύησεις πιο πολύ από αυτό που πρότεινε αρχικά το Συμβούλιο. Όποιο και να είναι λοιπόν το αποτέλεσμα, στηρίζω τροπολογία αυτή. Υπάρχουν και κάποιες άλλες τροπολογίες που αποσύρθηκαν κατά τα άλλα. Δεν βλέπω άλλες δυσκολίες, εκτός αν κάποιος θέλει κάτι να μου αναφέρει εδώ. Ξέρετε, εργαστήκαμε μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ήταν εύκολο να προετοιμάσουμε την ψηφοφορία σήμερα το πρωί. Θελήσαμε όμως να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ελπίζω μετά την ψηφοφορία να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Πραγματικά εργαστήκαμε ως τελευταία στιγμή και σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας για αυτές τις τελευταίες ε, αλλαγές. Σας ευχαριστώ κυρία Λάτφορτ. Καταλαβαίνω ότι προτείνεται εδώ και μια προφορική τροπολογία. Θέλετε να ψηφίσουμε γι' αυτό. Ή θα περιμένετε τη στιγμή που θα φτάσει η στιγμή να συζητήσουμε, δηλαδή για το 39. Ναι, ναι, όταν φτάσουμε στο 39... Αλλά πραγματικά, Πρόεδρε, όπως θέλετε, εγώ προτείνω όταν φτάσουμε στο σημείο αυτό να ψηφίσουμε για την προφορική τροπολογία και κατόπιν, ε, αν αυτό δεν περάσει, να πάμε στο κείμενο το αρχικό ή να πούμε ότι η τροπολογία 39 όπως έχει τροποποιηθεί και να την ψηφίσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν την ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρος. Είστε έτοιμοι. Ξεκινάμε με την τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 68 αποσύρεται. 69 υπέρ κατά εγκρίνεται 15 καταπίπτει 16 υπέρ κατά εγκρίνεται 17 υπέρ κατά εγκρίνεται 18 υπέρ κατά εγκρίνεται 19 υπέρ κατά εγκρίνεται 70 είναι γλωσσική δεν ψηφίζουμε συμβιβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά εγκρίνεται η 71 καταπίπτει, η 20 επίσης. Ψηφίζουμε την 72. Κατά. Εγκρίνεται. 74 καταπίπτει, 73 επίσης. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 21 καταπίπτει, 75 επίσης, 76. Ξεχωριστή ψηφοφορία για την 76. Όχι, καταπίπτει, συγγνώμη. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα του 76 υπέρ κατά εγκρίνεται να ελέγξουμε όχι δεν ελέγχουμε εγκρίνεται Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 23, 77 και 78 καταπίπτουν. 24 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται η καταπίπτει η 25, η 79, η 80, η 81. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 26, 82, καταπίπτουν. Ψηφίζουμε την 27 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 2983. Ψηφίζουμε την τροπολογία 84. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. 15 υπέρ, 26 κατά, 2 αποχές, απορρίπτεται. Ψηφοφορία για την τροπολογία 85. Είναι ίδια. Περνάμε στην 80. Ε, ε, συγγνώμη, στην 30. 30. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Απορρίπτεται η 30. Ελέγχουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 28 κατά. Απορρίπτεται η 30. Η 86 καταπίπτει. Η 86, όχι. Όχι, δεν καταπίπτει. Καταλαβαίνω, λέει ο πρόεδρος. 86, ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Για την 86 ψηφίζουμε. Τέλος. Υπέρ 25. Κατά 18. Εγκρίνεται η 86. 31. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 86 7. Κατά. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά εγκρίνεται. 36 ξεχωριστή. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά νομίζω ότι απορρίπτεται. στο τμήμα υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Ογδόντα οκτώ. Καταπίπτει. Ψηφίζουμε για την 88. Ψηφίζουμε. Ή δεν ψηφίζουμε. Ας ψηφίσουμε την 89 τότε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 90. Όχι. Κατά πίπτη. Αποσύρθηκε, συγγνώμη. 37. 37 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. 93 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα φτάσαμε στα εκτιμώντα, λαμβάνοντα υπόψη κτλ. 39, τροπολογία 39, υπέρ. Μα εδώ είναι που όπως θυμάστε υποβάλλω μια προφορική τροπολογία. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η προφορική τροπολογία αναφέρεται στο κείμενο της οδηγίας και λέμε ότι λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μία πρόταση και τα λοιπά. Δεν αναφερόμαστε δηλαδή στη νομική βάση. Υπέρ της προφορικής τροπολογίας ψηφίζουμε. Κατά εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά Εγκρίνεται. 40, 41, 42 καταπίπτουν. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Οι δύο καταπίπτει. Και τώρα ψηφίζουμε την 43 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε τη 44. Την 45 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 46. Όχι, όχι. Δεν την ψηφίζουμε. 47 υπέρ κατά νομίζω ότι εγκρίθηκε 48 Θέλετε να ελέγξουμε πια; Την 47. Ψηφίζουμε την 47. Αρχή της ψηφοφορίας. 47. «25 υπέρ 17 κατά». Εγκρίθηκε η 47. 48 υπέρ κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 9 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Η τρία καταπίπτει. Και ψηφίζουμε τώρα για τη 49 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 4 καταπίπτει. Ψηφίζουμε την 50. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 51. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 53 είναι ίδια, η 52 καταπίπτει, η 54 επίσης, η 6 επίσης. Ψηφίζουμε την 7, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 55 καταπίπτει. Συμβιβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 8 καταπίπτει. 56 υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε. Ηλεκτρονικά. Όχι. Εντάξει. Εγκρίθηκε. Η 9 τώρα. Υπέρ. Κατά. Η 10. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Συμβεβαστική τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Η 11 καταπίπτει και η 57 Ψηφίζουμε τη 12. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 58. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 59. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 60. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Με μια προφορική τροπολογία του ΕΛΚ. Κατά. Εγκρίνεται. 62. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 63 καταπίπτει. 64 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 65 είναι ίδια. 13 υπέρ της 13. Κατά εγκρίνεται. 66 καταπίπτει. Η 67 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. 27 υπέρ, 6 κατά. Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Λάτφορτ. Thank you. That concludes our work for the time being. Next. La próxima sesión es el 26. 26, 27, and 28. If, if there is no, we have concluded our work. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει τις ε, ψηφοφορίες για σήμερα. Αν δεν υπάρχει ε, κάτι άλλο, λίγη και συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 26 Απριλίου.